Μια κυρία που μας υποστήριζε πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Μπριγκίτ Στέλτσμποργκ, μας εγκαταλείπει. Μπαίνει σε σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου. Μπορείτε να σηκωθείτε. Κυρία,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 να τα παρουσιάσω. Καταρχάς έχω μια έκκληση να απευθύνω προς όλο το Κοινοβουλίο που αναφέρεται σε ένα κατεπήγον θέμα το οποίο θα ε, συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα για την κυρία Αμινά του Χαϊντάρ. Σήμερα το απόγευμα προβλέπεται κατεπήγον θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ζητώ την εμπιστοσύνη των συναδέλφων ε, για την ε, εξή διαδικασία. Κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό θα γνωρίζουν και δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε στην παρούσα φάση, αλλά το γνωρίζω και εγώ ότι λίγο, βρισκόμαστε λίγο πριν μία, μίας λύσης για την υπόθεση αυτή σήμερα, γιατί οι εκπρόσωποι και αρχηγοί κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζονται για την εξέβρεση μιας λύσης. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να διαγράψουμε αυτό το κατεπήγον θέμα από τα από την ημερήσια διατάξη σήμερα, γιατί κάθε περαιτέρω συζήτηση ε, νομίζω ότι θα παρεμποδίσει τις διπλωματικούς οδούς. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να διαγραφεί το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη, γιατί νομίζω ότι πιο πολύ θα παρεμποδίσουμε παρά θα βοηθήσουμε το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη έκκληση. Πρόεδρε, τη δεύτερη έκκληση θα την παρουσιάσω σε λίγο. Κύριε συνάδελφοι, δεν είμαι πεπισμένος ότι το θέμα αυτό μπορεί να συζητηθεί τώρα. Φοβούμαι ότι είναι αργά να κρίνουμε επί του τίματός σας αυτή τη στιγμή. Ήδη λάβαμε μία απόφαση επί του θέματος, άρα είναι δύσκολο για μένα να ξανανοίξω τη συζήτηση στο σημείο αυτό. Παρακαλώ, κύριε Ντόλου, πρόεδρε, υποστηρίζω την πρόταση του Μαρτίν Σούλτς. Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες. Μιλούμε για μια περίπτωση ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας. Προσπαθούμε να βρούμε μια πολιτική λύση. Νομίζω λοιπόν όταν, ότι όταν γίνεται προσπάθεια να βρεθεί πολιτική λύση δεν πρέπει να επιδεινώσουμε την κατάσταση. Ζητώ λοιπόν να αφήσουμε πρώτα να βρεθεί πολιτική λύση. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πόρτας, ο κύριος Πόρτας ήθελα να πω το εξή. Είναι πολύ σημαντική η διπλωματική δουλειά. Αλλά η αμυνά του Χαϊντάρ είναι στην 13η, 14η μέρα απεργίας πείνας στο νοσοκομείο. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε σε μια γυναίκα που αγωνίζεται για βασικά θεμελιώδη δικαιώματα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αγνοεί, την ξεχνάει. Ευχαριστώ. κυρίε και κύριοι. Μισό λεπτό. Βάση του άρθρου 140 του κανονισμού μπορούμε να ψηφίσουμε μια τέτοια πρόταση διότι υποβλήθηκε στην ουσία έτοιμα να φύγει ένα θέμα από την ημερήσια διάταξη. Το άρθρο 140 του κανονισμού επιτρέπει να γίνει ψηφοφορία επί του σημείου αυτού. Θα ήθελα να ζητήσω από το σώμα να μου πει ποιος θα μιλήσει υπέρ του αιτήματο και ποιος, ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ του αιτήματο. Ο κύριος Λόπες Αγκύρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως επικεφαλής της σοσιαλιστικής αντιπροσωπείας στο ε, Κοινοβούλιο θέλω να υποστηρίξω την άποψη του Προέδρου της ομάδας της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών της Ευρώπης που υποστήριξε και ο Πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρώτον, το Κοινοβούλιο αυτό σίγουρα εκφράζει την αλληλεγγύη την αλληλεγγύη του με την αμυνά του Χαϊντάρ και τον αγώνα της. Σε αυτές τις που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ζωή λόγω μια παρατεταμένη απεργία πείνα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, εκφράζουμε μια σωστή χειρονομία υποστηρίζοντα την εντατική διπλωματική δραστηριότητα που ε, πραγματοποιείται αυτέ τι μέρε με βάση την ε, ισπανική κυβέρνηση που είναι η κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αμυνά του Χαϊδάρ και είναι η κυβέρνηση μιας χώρας στην οποία πραγματοποιείται μια απεργία πείνας ενώ η ίδια η αμυνά του Χαϊντάρ είπε ότι δεν θα τελειώσει εάν δεν μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα της. Διακόπτει ο πρόεδρος. Υποστηρίζουμε λοιπόν την διπλωματική προσπάθεια που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε ένα ψήφισμα που θα μπορέσει να εμποδίσει την ε, εξέλιξη της κατάστασης και να αλλάξει διακόπτει ο πρόεδρος. Ποιος θέλει να μιλήσει κατά. Παρακαλώ. Θα σας πω γιατί η δική μου ε, ομάδα είναι κατά. Θεωρώ ότι δεν είναι ευτυχής η στιγμή που επιλέξαμε. Και όχι μόνο αυτό, δείχνει και έλλειψη σεβασμού προς όλες τις ε, πολιτικές ομάδες οι οποίες έχουν καταθέσει προτάσεις ψηφίσματος. Χθες συγκεκριμένα τρεις ώρες ε, συζητούσαμε το θέμα. Για να Πρέπει δηλαδή να αφήσουμε εκτός ε, αυτό το θέμα για να μην δοθεί προσοχή στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Εμείς προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ψήφισμα και το καταφέραμε. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα. Στη συνεδρίαση επίσης διαπραγματευθήκαμε κάποιες ε, διαφωνίες και αντιθέσεις. Δεν είναι λοιπόν σκόπιμο αυτό. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσει για αυτή την περίπτωση. Αν δεν το κάνει τώρα, ε, πότε θα το κάνει. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι σαφή η κατάσταση. Σα ευχαριστώ όλου. Κυρίες και κύριοι, θα ψηφίσουμε ποιος είναι υπέρ της υιοθέτησης της πρότασης. Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας. Επί της διαδικασίας. Διαδικαστικό, πρόεδρε. Ζήτω το λόγο δεν μου το δίνεται. Δεν είναι αληθές ότι το Κοινοβούλιο έλαβε θέση για την κυρία Χαϊντάρα. Δεν είναι αληθές. Σήμερα θα λάβει θέση. Σήμερα. Μετά από 33 μέρες απεργίας πείνας. Και μου λέτε ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε το θέμα σήμερα. Αυτό είναι ανήθικο. Πραγματικά ανήθικο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ψηφίζουμε. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. Άλλο διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για διαδικαστικό. Αυτό το κοινοβούλιο έχει μία σταθερή δέσμευση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έκανε μία πρόταση σήμερα το πρωί ο κύριος Σούλτς Εάν έχει στοιχεία και πληροφορίες σημαντικές σχετικά με την ε, υπόθεση Χαϊντάρ, ας μας τις διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες και να λάβουμε την απόφαση το μεσημέρι, πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Σούλτς, εδώ και πολλά έτη βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο και είμαι υπεύθυνο για τις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξ ονόματος της ομάδας μου και με μεγάλη προσοχή παρακολουθώ τα θέματα αυτά και θα ήθελα να πω ότι την προηγούμενη Κυριακή μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου επί ε, ώρες και μου δόθηκε η εντύπωση ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα η απεργία πείνα της κυρίας Χαϊντάρ να λάβει ένα τέλος και να εξευρεθεί λύση. Αν είχα την εντύπωση ότι με μια δημόσια δήλωση του Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του θέματος, θα είχα προβεί σε αυτή τη δήλωση, γιατί θεωρώ ότι σε τέτοιες σύνθετες διπλεωματικές υποθέσεις, η διακριτικότητα είναι η λύση του προβλήματος. Παρακαλώ τους συναδέλφους να συμβάλλουν με αυτή τη διακριτικότητα στη σωτηρία της γυναίκας αυτής. Αυτό είναι το έτοιμά μου. E, Κοιτάξτε, θα ήθελα να με προσέξετε ένα λεπτό. Δεν μπορούμε να παρατείνουμε εσάι την συζήτηση για το σημείο αυτό. Άλλος τελευταίος που ζήτησε το λόγο. Ο συνάδελφος από την θέση 92. Κύριε Ζαρμέρα, πρώτα απ' όλα εκπλήσωμε, διότι όπως είπε και η κυρία Μπιλμπάου πολύ σωστά, χθες είχαμε μία συζήτηση σχεδόν τρίωρη για αυτό το θέμα. Αν ο κύριο Σούλτ είχε πληροφορίε από την Κυριακή ότι έτσι είχαν τα πράγματα, έπρεπε να τα γνωρίζαμε τα στοιχεία αυτά χθε. Πρωτού καταλήξουμε στο ψήφισμα. Εάν δεν είναι έτσι τα πράγματα, χθε τι συζητήσει που είχαμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων και όπου καταλήξαμε σε συμβιβασμό, σε συμφωνία. Ακούστε, συμφωνήσαμε επί ενό κειμένου χθε. Δυστυχώ κάποια σχόλια εκτό μικροφών, Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε την ευθύνη να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα ώστε να γίνει γνωστή τουλάχιστον η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αμυνά ε, του ΧΑΙΔΑΡ. Δεν δέχομαι να μην γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Πρόεδρε, προφανώ υπάρχει διαφορά μεταξύ των μελών του σώματο. Είναι περίπλοκο το θέμα και υπάρχει σύγχυση. Θα ζητούσα να αναβάλουμε μέχρι τις 3 την ψηφοφορία, ούτως ώστε να γίνει μια συζήτηση μεταξύ ομάδων και κομμάτων και να λάβουμε υπόψη μας και να μάθουμε και τι έγινε επί τόπου. Ευχαριστώ. Uh, Κυρίες και κύριοι, συλλέξαμε και ακούσαμε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε σχηματίσει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα 140 του εσωτερικού μας κανονισμού θα ήθελα να θέσω σε ψηφοφορία το αίτημα του κυρίου Σούλτς καταρχάς για την διαγραφή από την ημερήσια διάταξη του συστήματος αυτού. Ποιος είναι υπέρ της διαγραφής παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ποιο είναι κατά. Δηλαδή θέλουν να παραμείνει το θέμα στην μερική διάταξη. Σας ευχαριστώ. Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασης ψηφοφορίας. 249 ψήφοι υπέρ, 163 κατά, 135 αποχές. Επομένως εγκρίνεται το αίτημα αυτό της διαδικασίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σούλτς για το δεύτερο διαδικαστικό. Πολύ λυπάμαι που σας ταλαιπωρώ, Πρόεδρε, και το υπόλοιπο Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, στον κατάλογο των ψηφοφοριών έχουμε την ψηφοφορία για την αρχή της επικουρικότητας. Ζητώ βάση του άρθρου 171 παράγραφος 4 του κανονισμού να μην γίνει ψηφοφορία, να αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι την επόμενη ρομέλη για το θέμα αυτό. και να ελέγξουμε την παρατακτότητα της, ε, του ψηφίσματος αυτού. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι οι αρχές της επικουρικότητας και του βασικού δικαίου είναι διασφαλισμένα. Δεν έχει νόημα όμως να το θέσουμε αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να πω και εξ ονόματος των Ιταλών συναδέλφων μου ρετά ότι η συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία είναι μια συζήτηση η οποία είναι Ιταλική, όχι Ευρωπαϊκή. Και συνάδελφοι, έτσι υπερασπιζόμαστε και προασπιζόμαστε την διαφορετικότητα και την πολυμορφία. Δεν έχει νόημα σε ένα τέτοιο ψήφισμα, δεν έχει νόημα σε ένα τέτοιο ψήφισμα να κατεβάσουμε τέτοιες προτάσεις τώρα. Πρόεδρε, πρόεδρε, πρόεδρε είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι ομάδες, ότι οι ομάδες λέω, οι οποίες είναι δημοκρατικές δεν γνωρίζουν το δημοκρατικό δικαίωμα ενός ομιλητή να μιλήσει. Σας παρακαλώ. Γι' αυτό ζητώ βάση του άρθρου 171 παραγράφου 4 την αναβολή της ψηφοφορίας για την επόμενη ολομέλεια και τον έλεγχο της παραδεκτότητας του ψηφίσματος καθώς και της ε, ψηφοφορίας του. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Έχω μια συγκεκριμένη πρόταση. Παρακαλώ κύριε Σούλτς, φορέστε τα ακουστικά σας για να με ακούσετε. Λοιπόν, έχω μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό το θέμα είναι στη δεύτερη ε, δέσμη ψηφοφοριών. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον προπολογισμό. Μπορείτε λοιπόν με την ησυχία σας να σκεφτείτε όλοι την πρόταση του κυρίου Σούλτς και να επανέλθουμε όταν θα έρθει η σειρά αυτού του θέματος, στη δεύτερη επαναλαμβάνω δέσμευση ψηφοφοριών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ψηφίζουμε τώρα επί του προϋπολογισμού. point of order. Κύριε Πόσελτ, διαδικαστικό έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομο. Ζητώ, επειδή διαγράψαμε το κατεπήγον θέμα και χτες ε, συζητήσαμε το χρόνο ομιλίας για τα καταπήγοντα και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, να μοιραστεί ο χρόνος ομιλίας που είχε προβλεφθεί για τη Δυτική Σεχάρα και τα άλλα δύο θέματα για να έχουμε αρκετό χρόνο για σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μία ώρα καταπήγοντα θέματα. Αυτό ήθελα μόνο να πω, Πρόεδρε. Ε, θα εξετάσουμε την πρότασή σας, κύριε Πόσελτ. Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε. Ψηφοφορία επί της εκθέσεως του κυρίου Μπέγκε.